έχουμε, αν δω, 3,38%. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι μόνο σημαντικό ρώσιμο το 20% σαν τις δαπάνες, ως άνωτη αύξηση, αλλά και τα 3 δις ως όριο. Τα, τα 2 δις, συγγνώμη. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο αυτά τα 2 δις θα υπερβληθούν με τον τρέχοντα προπολογισμό ή του χρόνου και νομίζω ότι ο υπεύθυνο ε, για την έκθεση του χρόνου θα πρέπει επίση να φροντίσει να μην υπερβληθεί το όριο των δύο δι. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό. Και θέλω να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων σε ό,τι αφορά και τις συνέπειες του Brexit. Αυτό που είναι σαφές είναι το εξή ε, ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ένα πακέτο το οποίο ενδεχομένω να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση μέχρι το 2020. Εκεί βρίσκονται στην παρούσα φάση διαπραγματεύσει. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι αν υπάρξει σκληρό Brexit από 1η Απριλίου του επόμενου έτου, μπορούν να αλλάξουν σημαντικά ορισμένε από τι συνθήκε αυτέ. Ποιε θα ήταν λοιπόν οι συνέπειε ενό σκληρού Brexit, κυρίω ό,τι αφορά και την εσωτερική κατάσταση στην ε, πολιτική ζωή της ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Σκοτία, δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει να εξέλιξεται η κατάσταση στην Ιρλανδία και μην σας πω, ότι δεν ξέρουμε και τι θα γίνει στο Γιβραλτάρ. Όλα αυτά λοιπόν ενδεχομένω να επηρεάσουν τη διαπραγματευτική μας ε, κατάσταση. Μπορεί να θέλουν να μείνουν μέχρι τι ευρωεκλογέ, μπορεί θεωρητικά να θέλουν να μείνουν μέχρι το 2020. Άρα οι διαπραγματεύσει πάντα θα πρέπει να προσαρμοστούν σε όλε αυτές τις εξελίξεις. Το θέμα της ευελιξίας ε, του προπολογισμού προφανώς είναι μεγάλο ζήτημα. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω ότι ποια είναι η άποψη των συναδέλφων. Ένα θέμα το οποίο, το οποίο πιστεύω ότι είναι θετικό ότι συζητιέται κάθε χρόνο είναι το επίδομα γενικών εξόδων. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι εφάπαξ ποσό κατά αποκοπήν. Και εδώ θα, θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη ευελιξία και η μέγιστη διαφάνεια. Είναι σαφές τι ποσό λαμβάνουμε. Και για μένα το καλύτερο λοιπόν θα ήταν αυτό. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, στα κρατημέλη υπάρχει ένα ποσό ε, θα για τα χιλιόμετρα που διασχίζει κανείς. Ε, δεν χρειάζεται να αποδεικνύουμε όμως σε κάθε περίπτωση τι αυτοκίνητο ε, οδηγάμε, τι καύσιμο και με λοιπά. Είναι φάπαξ το ποσό. Και όταν το υπερβούμε το άνοδο το όριο, πολύ απλά θα βάζουμε από την τσέπη μας μετά ο αξιωματούχος δηλαδή τα βάζει την τσέπη του. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ε, το πιο σωστό και το πιο σαφές για το επίδομα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της περσινές με τις οποίες ασχολήθηκα επισταμένως. Εξέτασα και την ε, ιστοσελίδα του κάθε βουλευτή και του Κοινοβουλίου για το πώς ε, μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθήσουμε και τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Εγώ τι έκανα. Έκανα ένα screenshot από κάθε homepage, από κάθε αρχική σελίδα του κάθε βουλευτή και του κοινοβουλίου, της ιστοσελίδα του κοινοβουλίου, να δούμε πώς ε, αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό του ποσού κατά αποκοπή και διαπίστωσα ότι κανένα βουλευτή ε, δεν ε, έδωσε πληροφορία για το τι κάνει με το ποσό αυτό κατά αποκοπή. Ίσως Μπορούμε να το αφήσουμε αυτό στην διακριτική ευχαίρεια του καθενό, αν κάποιον τον απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Και με χαρά θα πρέπει να σα πω ότι διαπίστωσα και την μπορώ να βελτιώσω και στη δική μου σελίδα. Τώρα, για το κόστο τη προεκλογική εκστρατεία. Πάντα αποτελεί αυτό μια πρόκληση, γιατί φυσικά το κόστος αυτό τίφεται και υποκριτήρια συμμόρφωσης. Ε, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Εδώ οι προδιαγραφέ ε, είναι πλέον αρκετά εκτεταμένε. Και φυσικά θέλουμε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων αυτών και το Κοινοβούλιο από ό,τι μας εξήγησε και ο Γενικό Διευθυντή, είναι καλά προετοιμασμένο και θα προσπαθήσει να βοηθήσει και να μας καλύψει με αντικειμενικό και καθαρό τρόπο μέχρι τις ευρωεκλογές. Έχουμε και τις πιστώσεις για ε, τα έξοδα και τις δαπάνες αναβαλαίωσης και εξυγχρονισμού των κτηρίων. Και εδώ και στο Στρασβούργο ε, έχουμε το θέμα της εξασφάλισης ε, των συνταξιβητικών δικαιωμάτων των βουλευτών και τίθεται για το θέμα της συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών και με την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Εδώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλές οι τροπολογίες που κατατέθηκαν για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σφιχτό προπολογισμό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εφαρμόσω και να υποστηρίξω όλες τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με μείωση της δαπάνης των χρημάτων των φορολογημένων και σε ό,τι αφορά τη μέγιστη, για παράδειγμα, το μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού κτλ. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε καλούς συμβιβασμούς. Γενικά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας πρότεινα να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και προηγουμένως ε, στη συνεδρίαση και κλεισμένα των θυρών. Να δώσουμε το λόγο πρώτα στους κοιότης. Είμαστε λίγο πιο νωρίς από ό,τι προβλεπόταν στο πρόγραμμα. Α, συγγνώμη, μάλλον έχουμε καθυστερήσει ενδεχομένω. Θα σας ε, ε, παρακαλέσω λοιπόν να μιλήσετε ένα λεπτό μόνο. Το λόγο λοιπόν, αν τον επιθυμεί, τον έχει η κυρία Καρτία Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο ένα λεπτό που μου δίνεται. Έχουμε ακούσει τον κύριο Ρουμπίχ πάρα πολλές φορές. Οι τροπολογίες μας στοχεύουν στη διατήρηση ε, του επίπεδου των τακτικών δαπανών κάτω από τον προϋπολογισμό, η αύξηση δηλαδή αυτών, και γενικά να είμαστε κάτω από τα δύο δις που υποτίθεται ότι είναι ο μαγικός αριθμός. Παρουσιάσαμε σειρά τροπολογιών για τα APAs, για τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, για τις αποστολές να είναι το ίδιο επίπεδο με τη γραμματεία ζητήσαμε από το Προεδρείο να αλλάξει τους κανόνες έτσι ώστε οι υπότροφοι που προσλαμβάνονται ε, να έχουν αξιοπρεπή μισθό, η όσοι κάνουν μαθητεία δηλαδή και στάζ, και να μπορούμε να έχουμε επαγγελματίες για τα διάφορα καθήκοντα. Για το Brexit τώρα. Όπως και να γίνει και ό,τι και να είναι, το ίδιο θα είναι για το Κοινοβούλιο. Οι Βρετανοί βουλευτές θα φύγουν, θα μας εγκαταλείψουν τη μέρα που θα τεθεί σε ισχύ. Επομένως αυτό μπορούμε να το ε, βάλουμε στον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να είναι εδώ ο κύριος Κολμέλο. Ο κύριος Άλλη τον είδαμε, αλλά δεν βλέπω να είναι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Ο κύριος Ντεπρέ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Το υπενθυμίσατε κι εσείς. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής για την ΑΛΤΕ. Ο κύριος Αλή όμως απουσιάζει και τον αντικαθιστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ προσοχή τα λόγια του συναδέλφου Ρούμπιχ και είπε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είπε ότι από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί κάποιες είναι θετικές. Εξαιρετικό το νέο αυτό, το βρίσκω. Εξαιρετική διατύπωση ότι κάποιες από αυτές που υποβάλαμε είναι εξαιρετικές. Ελπίζω και οι δικές μας έτσι να χαρακτηριστούν. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, με δύο λόγια. Σημειώνω τα λόγια του κυρίου Ρίμπιχ. Να μας τα διευκρινίσει όμως. Γενική αύξηση του προϋπολογισμού θέλει να είναι περιορισμένη στο επίπεδο του πληθωρισμού, σε γενικέ γραμμέ, επαναλαμβάνω, συνολικά. Καλά κατάλαβα, κύριε Ρουιμπίχ. Γνωρίζει μήπως ο κύριο Ρουιμπίχ ποιο ποσοστό θα πάρουμε ως πληθωρισμό για σημείο αναφορά. γιατί έχει μια μικρή σημασία. Τώρα, ως προς την Άλτε, τη δική μου πολιτική ομάδα, και το είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε κάτω από τα 2 δις ευρώ. Είμαστε σε έτος προεκλογικής εκστρατείας και μέρος της κοινή γνώμης και των μέσων επικοινωνίας. Υπάρχουν πάρα πολλές ευαισθησίες σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση του προπολογισμού. Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι όταν αυξάνουμε τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου τα βάζουμε στην τσέπη μας. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κάναμε κάποια σχέδια για εξοικονομήσεις και θα ήθελα να επιμείνω σε κάποια. Καταρχάς, σε προηγούμενη συνεδρίαση είχα αναρωτηθεί πράγματι χρειάζονται αυτές οι διατευθετήσεις για τα κτίρια. Όταν περπατώ και περιδιαβαίνω το 15ο όροφο, εκεί που είναι το γραφείο μου, Βλέπω το 12ο, τον 8ο και λέω, μα ποιο τα αποφάσισε και γιατί είναι επίγον και ποιο είναι ο στόχος και γιατί τα κάνουμε αυτά. Έχει νόημα αυτό το πράγμα. Και άλλε αποφάσεις έχουν ληφθεί που είναι πολύ ιδιαίτερε. Ίσως με θεωρείτε παλαιομοδίτικο που τα λέω αυτά. Αλλά αποφασίσα να, να έχουμε webcam και παντού και ποιο το αποφάσισε αυτό και γιατί, σε ποιον προορίζεται, να μοιράσουμε και επίση και κράνη νομίζω κάπου είδα στον προπολογισμό, γιατί. Δηλαδή, σε θέματα εξοπλισμού και εργασιών στα κτίρια ε, δεν τεκμηριώνονται αυτά, δεν δικαιολογούνται. Νομίζω ότι χωρίς καμία δυσκολία <laughs> μπορεί κανείς να προσαρμόσει τον προϋπολογισμό χωρίς να έχει καμία δυσκολία και να μην ξεπεράσει τα δύο Δύο είναι οι ιδέες που θα ήθελα. Α, έχω μόνο ένα λεπτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν είμαι υπέρ ε, ε, κατά, του καταποκοπήν ποσού για τις γενικές δαπάνες. το 122 δεν το συμφωνώ με αυτό για την κοινοβουλευτική βοήθεια και τους βοηθούς. Αυτά. Συνολικά είναι τα σχόλια για την ε, εκ μέρους πολιτικής μου ομάδας και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είχα ένα λεπτό μόνο στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Να δούμε τι μας... Ε, ποια είναι η άποψή σας. Ο επόμενος λοιπόν ε, στην σειρά είναι ο κ. Θέραντ. Ευχαριστώ. Σε ένα λεπτό να πάω τα πιο σημαντικά. Είμαι αισιόδοξο και χαρούμενος που είμαι σκιώδης ε, τον κύριο Ρούμπιχ, την κυρία Ρούμπιχ και στο πώς αντιμετωπίζει τις τροπολογίες, μερικές εκ των οποίων ήταν πραγματικά πολύ ριζοσπαστικέ από τις πράσινους. Ε, να τονίσω τρία βασικά ζητήματα, τα οποία ενδεχομένω μπορεί να βελτιωθούν, επειδή έχονται βελτιώσεις. Σε ό,τι αφορά την πολιτική, ε, για τα κτίρια, δεν είμαστε μηχανικοί, αλλά ο κ. Ντεπρέ τουλάχιστον έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κτιριών. Να υποστηρίξω λοιπόν ε, την προσέγγιση του σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κτιριών και να δούμε αν υπάρχει ευκαιρία να προβλεφθούν σωστά έργα συντήρησης όποτε χρειαστεί, όχι μόνο το 2019. Είναι λες και το απερχόμενο κοινοβούλιο αγνοεί τις ανάγκες αυτές, τις οποίες τις φορτώνει στις πλάτες του μελλοντικού κοινοβουλίου. Ίσως να μην είναι η καλύτερη πολιτική αυτή. Δεύτερον, να αναφέρω πάλι αυτό το ευαίσθητο ζήτημα του εθελούσιου ταμείου συνταξιευδότησης και να ζητήσω μια τροποποίηση αυτού, αν όχι απόσυρση. Και τρίτον, η πιστοποιημένη βοηθή και το θέμα της συνταξιοδότησης, του Ταμείου Συνταξιοδότησης τους. Αν ε, το λύσουμε αυτό το θέμα θα μας είναι αιώνια ευγνώμονη η βοηθή αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάνη. Ευχαριστώ πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε χρόνο να συζητάμε αυτό το θέμα σε τέτοιου τύπου συνεδριάσεις ε, εισηγητών. Να είμαστε, ναι, όντως, να μείνουμε κάτω από τα δύο δισεκατομμύρια, αλλά γιατί το βασικό θέμα είναι να, να χρησιμοποιήσουμε με τρόπο έξυπνο τα λεφτά των φορολογουμένων. Κάναμε κάποιες προτάσεις για περικοπές δαπανών. Υπάρχουν πολλές γραμμές του προπολογισμού που μπορούμε να περικόψουμε. Δεν συμφωνώ επομένω με τον κύριο Ντεπρέ για, το τι πρέπει να, για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε περικοπές. Ε, το βασικό είναι να έχουμε λεφτά και να υπάρχει ε, διαφάνεια. Για τα γενικά έξοδα και τις αποζημιώσεις ε, των γενικών εξόδων μπορούμε να κάνουμε μια έξυπνη δουλειά να πάρουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο ε, της δικής μας αποζημίωσης και τα έξοδα να αποζημιώνονται όταν, γίνεται, όταν καταβάλλεται η αίτηση. Ε, είναι ένας απλός τρόπος αυτός. Ε, τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε όταν ε, τα πούμε μεταξύ μας, μεταξύ σκιωδών. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριο Χαουαρτίδα μας ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συγκρίσεις εντός του Κοινοβουλίου, είναι, όπως ανέφερε ο κύριος Ζούμπικ, είναι χρήσιμες και μπορούμε να κάνουμε και συγκρίσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, με κάθε αναλογικότητα βέβαια. Ε, πάντως, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να χαρτογραφήσουμε τις ε, εξοικονομήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε αν είχαμε μία έδρα μόνο. Εάν ε, είναι σοβαρό ο κ. Μακχόν ότι θέλει να αλλάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω να συμφωνήσει ε, στην απαραίτητη αλλαγή τη συνθήκη για της, με σκοπό την αλλαγή τη έδρα. Καλό και άγιο να λέμε ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε τα λεφτά των φορολογουμένων. Προφανώς με υπέρ ε, και προφανώς μπορεί να κάνει κανείς ε, κάποιες ε, εξοικονομήσεις, αλλά πρέπει να δίδονται και οι απαραίτητοι πόροι όταν χρειάζονται. Και ένα από τα βασικά που συνέβη σαν στο Κοινοβούλιο όσοι ήμουν εγώ εδώ, που δεν ήταν πολλά χρόνια, είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό θέμα της ε, παρενόχλησης και σεξουαλική ε, σεξουαλικής παρενόχλησης. Και αν θέλουμε να τιμήσουμε το προσωπικό που δουλεύει εδώ, θα πρέπει ε, να δώσουμε τα απαραίτητα κονδύλια ε, και να δει ο κόσμος ότι τα διαθέτουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ε, κύριε Ντεπρέ, έχω να σας πω κάτι για τα θέματα τα τεχνολογικά. Ναι, ίσως έχουν νόημα κάποια από τα πράγματα που είπατε, αλλά προσοχή από τις ψευδοοικονομίες. Γιατί εάν χρησιμοποιούμε εκτεταμένα το software, μπορεί να ε, είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι, να εκτεθούμε πολύ περισσότερο. Ε, μην ξεχνάτε ότι ε, δεν πρέπει απλώς να λέμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό μόνο για να δείξουμε ότι το κάνουμε. Θα πρέπει να δουλεύει σωστά το περιβάλλον ας πούμε, το, της πληροφορικής. Ε, να μην κάνουμε δηλαδή εξοικονομήσεις για τις εξοικονομήσεις, αλλά ε, εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ. Δεν ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Κύριε Ρούμπιχ, αν θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια εκτελεκτικά, έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω καταρχά του συναδέλφου ε, για τις προτάσεις τους ε, και να σας ε, διαβεβαιώσω ότι θα κρατήσω αυτή την σκληρή στάση και στο Προεδρείο και στις τριμερείς διαλόγους ε, σε ό,τι αφορά τις οικονομίες και τις περικοπές και προσβλέπω στη διαπραγματεύση γιατί πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια εντούλη ιδιαίτερα πριν από τις ευρωεκλογέ να δαπανίσουμε με το πιο σωστό και οικονομικό τρόπο τους ε, πόρους και τις, ε, τα χρήματα του φορολογουμένου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τις προτάσεις σας. ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Νομοδότηση του κυρίου Άλλη για την Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Έχετε το λόγο κύριε Άλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ρόλος της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός γιατί εγγυάται την ασφάλεια των τροφίμων για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί εξαρτώνται από τη φύση και είναι οι βασικοί προστάτες του περιβάλλοντος. 6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ασχολούνται με τη γεωργία σήμερα και με τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων. Οι γεωργικές και δασοκομικές περιοχές, οι απομοκρισμένες, δεν χρησιμεύουν μόνο στην παραγωγή των τροφίμων, αλλά κατοικούνται από Ευρωπαίους πολίτες, είναι χώροι και περιοχές αναψυχής και τουριστικών δραστηριοτήτων. Έχοντας αυτά υπόψη, θέλουμε η ανακοίνωση για το μέλλον των τροφίμων και της ε, γεωργίας να εξεταστεί από την Επιτροπή Άγκρη για να πετύχουμε τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής να έχουμε, πρέπει να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του του δημοσιονομικού πλαισίου, να εξυγχρονίσουμε και να πλουστεύσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί ότι η λειτουργία του οικονομικού ελέγχου, του ε, οι έλεγχοι εκ των υστέρων και εκ των προτέρων θα γίνονται με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες συνθήκες σε όλα τα κράτη-μέλη. Και τρίτον, να γίνει κατανομή, δίκαιη κατανομή μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων, μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να μειωθούν οι αποκλήσεις ε, μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών και να δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στηρίζουμε όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και στο να βελτιωθεί η κατάσταση με τον ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να δούμε κατά πόσο ε, θέλει κανένα συνάδελφος να πάρει το λόγο. Α, μάλιστα. Ο κ. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλή για την έκθεσή του. Τους γενικούς προσανατολισμούς τους συμμερίζομαι, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανάγκη να εγγυηθούμε μια μελλοντική κάπο που θα έχει στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, τις νέες γεωργικές πρακτικές με, ε, με καλύτερο, καλύτερη χρήση της, του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, ε, με στήριξη το, της απασχόλησης και ειδικά των νέων. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να διευκρινιστεί γιατί θα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτόν τον ορισμό για να αμφισβητήσουμε την ε, καταλληλότητα των, ε, της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής για την ε, υπαίθρου της Ευρώπης, που δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε ποσοτικά και βραχυπρόθεσμα στοιχεία. Πολλοί εδώ ανησυχούμε για το νέο, το New Deal, το μοντέλο της Κομισιόν, δεν θέλουμε μια επανεθνικοποίηση τη της ΚΑΠ ε, ή στρεβλώσει από τα κράτη-μέλη. Τα καθαρά δημοσιονομικά στοιχεία της νομοδότησης ε, θα ήθελα να τα συμπληρώσουμε με τα εξή. Καταρχάς, μια ΚΑΠ η οποία όντως θα κρατηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο, στο μελλοντικό πουδουπού, ακόμα και όταν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, το σημερινό σύστημα επιδοτήσεων ε, δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί με χρηματοδοτικά άλλα εργαλεία. Οι άμεσες πληρωμές ε, δημιουργούν ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και ενισχύουν την ενιαία αγορά ε, μειώνοντας τις τρευλώσεις του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να βρούμε και τα νέα εργαλεία τα οποία θα μειώσουν την αστάθεια των τιμών και να αυξήσουμε την χρηματοδότηση των, προ... των προαιρετικών προγραμμάτων, ειδικά για τα πιο απομακρυσμένα εδάφη, αλλά και εκείνα που έχουν φυσικά προβλήματα ε, φυσικές δυσκολίες. Ε, τελευταίο σημείο, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις συνέργειες ε, ανάμεσα στην ε, υποδοχή των μεταναστών και στην ανάπτυξη των εδαφών της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί εφόσον το επιθυμεί. Thank you, Chairman. I think I can be very brief. Uh, Ευχαριστώ. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομο. Η έκθεση, Καθώ και το ψήφισμα των τελευταίων εβδομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτει διάφορα σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά το μέλλον τη ΚΑΠ. Δεν πρέπει να αναφέρω όλα αυτά τα στοιχεία ξανά. Θέλω να σα διαβεβαιώσω, ε, και όλα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζοντα τι προτάσει οι οποίε θα βγουν στις 2 ε, και στις 29 Μαΐου ε, εξετάζουν πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ναι, ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δευθυντά. Έτσι ολοκληρώνεται το σημείο αυτό στην ημερήσια διατάξη. Θα ήθελα να σα υποδείξω ότι σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα βρισκόμαστε σε διπλή δύσκολη κατάσταση. Από τη μία ε, έχουμε Του συναδελφού τη Επιτροπή Γεωργία που μα ενημέρωσαν πολύ καθυστερημένα και από την άλλη έχουμε και πράσινη εβδομάδα ενώπιον μα. Άρα οι τροπολογίε για την έκθεση του κ. Άλλη θα ληφθούν υπόψη μόνο στα αγγλικά. Είναι πραγματικά λυπηρό και απευκταίο, αλλά δεν βλέπω άλλη δυνατότητα αν θέλουμε να έχουμε κάποια επιρροή. Άρα προθεσμία είναι 28, 28 Μαρτίου. Και να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το 18, για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Ο εισηγητής είναι ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντος. Το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης, ε, το οποίο εκφράζει την ε, αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, για να επιλύσουμε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ε, λόγω κλιματικής αλλαγής ή λόγω άλλων λόγων, χρειάζεται να ενισχύσουμε αυτό το Ταμείο. Ε, με 500, το οποίο φτάνει στα 550 ε, εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει όμως το επόμενο που δουπού να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ μετά το 2020 λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κρατός μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να μην χρησιμοποιεί ε, τα κονδύλια των διορθωτικών ταμείων για την πρόληψη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προλάβουν παρά να διορθώνουν, παρά να θεραπεύουν όπως λέμε. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ μιλάμε για 104 εκατομμύρια, ε, ούτως ώστε η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία και η Ελλάδα στην περίπτωση ε, να μπορέσουν να στηριχθούν. Στην Πορτογαλία και στην Ισπανία έγιναν πυρκαγιές. Στη Γουαδελούπη, στο Σαμαχτά, Είχαμε επίσης της Γαλλίας είχαμε τυφώνες και στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολύ ισχυρού σεισμούς. 50,6 εκατομμύρια ευρώ ε, στην Πορτογαλία. Είχαμε πάνω από 1,4 ε, δις και χάσανε τη ζωή τους πάνω από 100 άτομα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτή πρέπει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Αυτός θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος. Γι' αυτό λοιπόν τονίζουμε την πρόληψη. Ε, για τη Γαλλία ε, έχουμε πάνω από ένα δις ε, ζημιές, 3,2 για τη Γαλλικία και ε, για την Ελλάδα η βοήθεια πάει στην, ε, στο νησί της Λέσβου. Μιλάμε για αλλαγές του προϋπολογισμού, ένα διορθωτικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το Ταμείο είναι ειδικό εργαλείο. Στην έκθεση εγώ ζητάω να υπάρξει ταχύτητα, υπάρχουν ε, κρατη που αυτά τα κράτη-μέλη χρειάστηκαν, ή κάποια τουλάχιστον από αυτά τα κρατη χρειάστηκαν χρόνο για να υποβάλουν τι αιτήσει. Τώρα θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και θα πρέπει να ψηφίσουμε στο Μάιο στην Ολομέλεια. Ε, και συνεχεία πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο το θέμα. Ε, Ούτω ώστε το χρήμα αυτό να φτάσει το στενότερο δυνατόν στι περιοχέ αυτέ. Ζητάμε διαφάνεια, ε, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στην εφαρμογή των, στην χρησιμοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου ε, για αυτές τις ε, περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές ε, καταστροφές. Ε, θα πρέπει να, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να κάνουν αναπρογραμματισμό για να προσθέσουν κονδύλια από τα διαρθωτικά ταμεία στις, προκειμένου να δοθούν στους πληθυσμούς αυτούς που επλήγησαν για να, και για να αποκαταστήσουν την οικονομία των πληγισών αυτών περιοχών και να ε, αποκαταστήσουν ας πούμε και την πολιτιστική κληρονομιά ή το φυσικό τοπίο κτλ. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει την τροποποίηση των ε, συμφωνιών εταιρική σχέση για να γίνει αυτή, αυτός ο αναπρογραμματισμός από τα κράτη-μέλη. Το ζήτησαν αυτό τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εγκριθεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή, αυτός ο επαναπραγματισμός επαναπρογραμματισμό είναι πάρα πολύ σημαντισμό και θα πρέπει ε, να συμπεριλαμβάνει και την πρόληψη, ούτως ώστε οι προβληματικές περιοχές να εντοπίζονται γρήγορα και σε αυτές τις περιοχές να γίνει το δύναμη, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν αυτές οι τραγωδίες και για να μην ξαναχαθούν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις περιοχές. Φυσικά, Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, καταστροφές που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά τουλάχιστον τις καταστροφικές επιπτώσεις να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις περιορίσουμε. Στις 27 Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Το Μάιο, όπως σας είπα, θα πρέπει να εγκρίνουμε στην Ολομέλεια αυτή την έκθεση επομένως αυτή η κινητοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Αλληλεγγύης που δείχνει και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις χώρες αυτές και που είναι στην τελική ε, ένα, μια σταγόνα ας πούμε ε, στην, στον ωκεανό αυτών των χρημάτων που θα χρειαστεί για να διορθωθούν οι ζημιές των τραγωδιών. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει η κυρία Γετενμάκη, τον εισηγητή, τον κύριο Φερναντές. Πολλά είναι τα πλέον εκτίματα που αποκομίζει κανείς στα θέματα πολιτικής προστασίας εάν συνεργάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλο και περισσότερες είναι οι φυσικές καταστροφές που σημειώνονται και μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση πολύ περισσότερο στο μέλλον, αφού δυστυχώς συνεχίζει ακάθεκτο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Συγγνώμη όμως, θα ήθελα να παρέμβω για κάποιο άλλο ζήτημα. Μιλούσατε για άλλο θέμα, μάλιστα. Ο κύριος Ντονάνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για αυτή την ε, απόφαση για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, για τις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και άλλες. Συμπάσχουμε με τις οικογένειες και τους οικείους ε, των θυμάτων. Συμφωνώ με τα λεγόμενα του κυρίου Φερναντές και κυρίως συμφωνώ ε, με το θέμα της πρόληψης. Θα υπερψηφίσουμε τις προτάσεις του και θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ζητάει κάποιος άλλος το λόγο από ό,τι φαίνεται. Για το θέμα αυτό, καταληκτική προθεσμία υποβολής λογιών είναι 27 Μαρτίου. Επομένως, περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμός 1, στο γενικό προϋπολογισμό του 18. Ο κύριος Μούρεσαν δεν μπορεί να είναι εδώ και έχει το λόγο ο κύριος Φερναντές γιατί είναι ο συντονιστής του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι ο πρώτος ε, διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2018. Συνοδεύει την ε, πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης ε, της ΕΕ που μόλις τώρα παρουσίασε. Μιλούμε για 141 εκατομμύρια ευρώ για 1,41 εκατομμύρια ευρώ. Καταληκτική προθεσμία είναι 28 Μαρτίου για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 16-17 Μαΐου στην Επιτροπή για τον προϋπολογισμό. Και προτείνω την έγκριση αυτής της διόρθωσης του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Θέλει το λόγο. Όχι, από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 27 Μαρτίου, είπατε 28 ή κάνω λάθος. Αν θέλετε να είστε σίγουροι, μέχρι τις 27. Και έτσι διεκπαιρεώνουμε και το σημείο 19 και περνάμε και πάλι στον ε, Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες για τον ε, Μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ένα αποθεματικό πόρων και μέσων για να μπορεί να βοηθήσει όταν σημειώνονται φυσικές καταστροφές. Όχι μόνο πυρκαγιές αλλά και σεισμοί, περίοδοι ξηρασίας, τρομοκρατικές επιθέσεις, πλημμύρες, και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει ένα αποθεματικό και να το αξιοποιεί, να το χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το αποθεματικό παρουσιάζει το εξής πλεονέκτημα, ότι μπορεί να δημιουργήσει αποταμιεύσεις και όπως είναι η περίπτωση της ε, καταπολέμησης των πυρκαγιών. Με λιγότερους συγκεντρωμένους πόρους καταφέραμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο βεληνικές, δηλαδή να, να, να, στοχεύσουμε σε περισσότερη βοήθεια. 15 αεροσκάφη κατασβεστικά που τα διαχειρίζεται κάποιο σε κεντρικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματικά από 50 αεροσκάφη τα οποία είναι κατακαιρματισμένα και διασπαρμένα στα, στα μέλη. Η διαχείρισή τους δηλαδή και η διοίκησή τους και έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες τέτοιων φαινομένων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Και τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής θα επιδεινώνονται. Οι ακραίες καιρικέ συνθήκες είναι όλο και πιο συνήθεις. Πρέπει όλοι να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί. Δεν αφαιρούμε αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη, όμως αυτός ο μηχανισμός πολιτικός, πολιτικής προστασίας είναι απαραίτητος μηχανισμός ε, ε, επίδειξη αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα το αποθεματικό αυτό, το εθελοντικό, είναι σημαντικό να μπορεί να αυξάνεται, να αυξηθεί. Και ελπίζω ότι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρόλο που είναι εθελοντικό αυτό, ότι θα είναι σε θέση να αυξηθεί. Τώρα, ως προς αυτό το συγκεκριμένο αποθεματικό μέσων, υλικών μέσων, για την περίοδο 2018-2020, προτείνεται αύξηση 280 εκατομμύρια ευρώ στην πρικοδότηση, στα μέσα που δίδονται. Και αυτό είναι καινοτομία, γιατί οι νέες προτεραιότητες πρέπει να έχουν επιπρόσθετους πόρους. Και γι' αυτό το λόγο η πρότασή μου η πρότασή μας από πλευράς προϋπολογισμού για αυτό το μηχανισμό πολιτικής προστασίας είναι να έχουμε αυτή την ποσότητα των χρημάτων, αλλά να μην τα πάρουμε από κάπου για να τα βάλουμε κάπου αλλού. Αυτά τα 80 εκατομμύρια να μην σημαίνει ότι θα τα στερηθούν άλλες σημαντικές πολιτικές για να τροφοδοτηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Όχι. Να χρησιμοποιήσουμε ε, εργαλεία ευελιξίας και να έχουμε νέα κονδύλια, φρέσκο χρήμα, να μην επανακατευθύνουμε υφιστάμενα χρήματα. Επομένως αυτά τα 280 εκατομμύρια ευρώ να είναι επιπρόσθετα και να χρηματοδοτήσουν αυτό το εργαλείο ευελιξίας. Θα δούμε τώρα εάν η αλληλεγγύη την οποία υποτίθεται τόσο θέλει το Συμβούλιο, αν θα την εφαρμόσει και στην πράξη, αν θα υιοθετήσει Προτάσει στην πράξη. Γιατί τι συμβαίνει στο Συμβούλιο, λένε τα μεγάλα τους λόγια και μετά όταν ε, έρθει η ώρα της πράξης <laughs> τελικά κάνουν τα αντίθετα. Η αλληλεγγύη δεν είναι κάτι που αναφέρει απλά κανείς, είναι κάτι που το κάνει, το πράττει. Πρέπει να δείξουμε ότι αυτά τα 280 εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετων χρημάτων για αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία που μιλούμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής να το αποδείξει και το Συμβούλιο ότι τη θέλει αυτή την αλληλεγγύη, την εστερνίζεται, την εφαρμόζει και είναι υπέρ του να δώσει αυτά τα επιπρόσθετα 280 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την προτεραιότητα, η οποία είναι συμπληρωματική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, βλέπω να θέλει να πάρει το λόγο κάποιο και ο Γι' αυτό λοιπόν ε, να δώσω το λόγο στου υπόλοιπου ομιλητέ, η κυρία Γετεμάκη. Και με μικρόφωνο, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπώ. Τώρα που είμαι στο σωστό σημείο της ημερησίας διάταξης, να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάντες για το σχέδιο γνωμοδότησης να σας πω ότι πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που μπορεί κανείς να αποκομίσει από την ευρωπαϊκή συνεργασία ε, στον τομέα της πολιτικής προστασίας και δυστυχώς ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε όλο και περισσότερες φυσικές καταστροφές. Να είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι. Το σημείο εκκίνησης βεβαίως θα πρέπει να είναι η ε, ευθύνη στα κράτη-μέλη οι εθνικές αρχές πρέπει να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις και είναι και ο πιο γρήγορος τρόπος για τη διάσωση, για την έρευνα και διάσωση. Αν πρέπει κανείς να περιμένει βοήθεια να έρθει από την απέναντι πλευρά της Ευρώπης, αυτό χρειάζεται χρόνος και στην περίπτωση των πυρκαγιών ίσως εξαπλωθούν πάρα πολύ μέχρι να έρθει η ξένη βοήθεια και θα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν αυτές οι πυρκαγιέ αν ε, χρειαστεί να περάσουν 5-6 μέρες μέχρι να έρθει βοήθεια από αλλού. Είμαι υπέρ της ε, ε, ε, αναδιάταξης και εκ νέου ανάπτυξης σπόρων, το redeployment, δηλαδή να πάρουμε πόρους από κάπου που δεν χρειάζονται και να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν εκεί όπου χρειάζονται. Είναι προγράμματα που έχουν υιοθετηθεί πολύ καλά και έχουν υψηλό ποσοστό απορροφησιμότητας κονδυλίων και συμφωνώ με αυτά. Όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε χαλεπούς καιρούς με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με το υπάρχει κενό στον προϋπολογισμό αφού φεύγουν οι Βρετανοί πρέπει να βρούμε αντισταθμίσεις να προσδιορίσουμε τις γραμμές του προϋπολογισμού που δεν είναι και τόσο επιτυχημένες με όσο τον καλύτερο τρόπο. Προτείνω λοιπόν να προετοιμαστούμε και να έχουμε αυτή την ευκαιρία να ασκήσουμε μια κάποια να σκηθούμε στη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν γίνεται συνεχώς αυτό το Νίκο να ζητούμε συνεχώς όλο και περισσότερα χρήματα. Να ζητήσουμε redeployment λοιπόν, ε, ανάπτυξη πόρων ε, σε κάποιους τομείς τους οποίους θα απορροφήσουμε από τομείς που υστερούν. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε περίπτωση η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί με τη δημιουργία και την εδραίωση αυτού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Στην Επιτροπή μας όμως δεν μιλούμε για την ουσία, μιλούμε για τα λεφτά. Εμείς λοιπόν ως σοσιαλιστές είμαστε πάντοτε υπέρ κάθε νέου εργαλείου, κάθε νέας πολιτικής και υπέρ του επιχειρήματος ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα νέο πράγμα πρέπει να έχει και νέα χρήματα. Λέει η κυρία Γετενμάκη, μα δεν μπορείτε να ζητάτε συνεχώ λεφτά. Απαντώ στην κυρία Γετενμάκη, αφού κάθε μέρα κάνουμε κάτι καινούριο, πρέπει να βρούμε καινούργια λεφτά. Δεν έχει νόημα να πάρουμε από τα προηγούμενα. Δηλαδή πρέπει για να φτιάξουμε ένα νέο πράγμα πολιτικής προστασίας να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να κόψουμε π.χ. από τις υποτροφίες Εράσμους που είναι τόσο επιτυχημένο πρόγραμμα. Κάθε φορά λοιπόν που δημιουργούμε κάτι νέο και διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής και χρησιμοποιούμε νέους πόρου, τότε πρέπει να βρούμε νέους πόρου. ιδαλλιώ ε, προχωρούμε ένα βήμα μπροστά στην καινούργια πολιτική και πάμε ένα βήμα πίσω στην παλιά. Δεν έχει νόημα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κανεί άλλο το λόγο. Να καλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο για να τοποθετηθεί. Αν ε, επιθυμείτε. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξη τη πρόταση και τα υπόλοιπα μέλη, του υπόλοιπου βουλευτέ που πήραν το λόγο. Να θίξω ένα θέμα μόνο, το θέμα τη ε, εκ νέου των πόρων. Νομίζω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κινείται σε μεγάλο βαθμό προς αυτά τα οποία ζήτησε ο εισηγητή. Αυτό που προτείνουμε είναι 90% καινούριο χρήμα, φρέσκο χρήμα σε ό,τι αφορά τη χρήση του εργαλείου ευελιξίας και μόνο 12% εκ νέου χρήση πόρων. Νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό κινείται προ την κατεύθυνση των όσων ζητάει ο εισηγητή. Σε ό,τι αφορά τι γραμμέ του προπολογισμού που ζητήσαμε, σε ό,τι αφορά τι ε, εκ νέου χρήσει αυτέ, κυρίω πρόκειται για τα θέματα ε, εργαλείων δικαιοσύνη και τέτοιων δικαιωμάτων, όπου εδώ δυστυχώ έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια μια χαμηλότερη απορρόφηση. Άρα δεν είναι ότι δεν έγινε σοβαρή και ενδελεχής εξέταση. Πιστεύουμε ότι με αυτή την περιορισμένη πρόταση αναδιανομής των πόρων θα υπάρξει ακόμα δυνατότητα ευελιξίας τα 2019 και 2020 για να μπορέσει να διασφαλιστεί η συνέχιση των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα είμαστε λίγο γρήγοροι. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας. Θα μπορούσε να έχει μιλήσει και λίγο παραπάνω ο κύριος τεπρέ. Τώρα ζήτησε το λόγο ο σκιώδης των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Βόλκαν. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Και συγγνώμη που καθυστέρησα, κύριε εισηγητή. Έχει Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχέδιο της γνωμοδότησης, την οποία έχει υποστηρίσει σε μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό για τις καταστροφές, ε, το μηχανισμό αλληλεγγύης, το θεωρώ πολύ σωστό, γιατί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπάρξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την πρόληψη καταστροφών. Το 2013 ήταν πολλά τραγικές ε, καταστροφές όπου και η συνεργασία δεν λειτουργήσε με το βαλτιστό τρόπο. Πιστεύω ότι είναι σωστή η αρχή. Ωστόσο στην πράξη έχουμε κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της συλλογική ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της δημιουργίας του ειδικού το οποίο θα είναι υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει κάποια αβεβαιότητα και ανασφάλεια στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το συντονισμό τη αντιμετώπιση κρίση, ε, κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα στο οικονομικό σκέλο ε, για το 2014 με 2020. Σύμφωνα ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μόνο το εργαλείο αλληλεγγύης και ευελιξίας και λοιπόν το θέμα το οποίο θα πετυχαίνουμε καινούριου στόχους χωρίς να φέρουμε πόρους από προηγούμενα προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να μην υπάρχει αδιανομή πόρων από τα κεφάλαια 3, 4 και 5. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, προστασίας δεν αποκλείει την ανάγκη πρόληψης. Την τονίζει ακόμα περισσότερο και αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα η αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Άρα η δημιουργία ενός συγκεκριμένου αποθεματικού είναι ένα συμπλήρωμα, κάτι το επιπρόσθετο, ένας επιπρόσθετος πόρος για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη ε, αν συμβεί μια φυσική καταστροφή, μια περκαγιά, ένα σεισμός, μια πλημμύρα, κάτι το τρομερό ή και τρομοκρατική επίθεση. Επομένως είναι επιπρόσθετα μέσα, επι, επαναλαμβάνω, που, δίνουν τη δυνατότητα να σωθούν ζωές. Και είναι μικρή η συνεισφορά των κρατών μελών και είναι και θελούσια. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε για να δρομολογηθεί αυτός ο μηχανισμός το συντομότερο, το γρηγορότερο. Βεβαίως η απόφαση πρέπει να ληφθεί όσο να τον πιο νωρίς, άλλο θέμα αυτό. Κατά την άποψή μου όμως αυτά τα 280 εκατομμύρια ευρώ για το 2018 έως και το 2020 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί αυτό το αποθεματικό και να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι που θα σώσουν ζωές είναι μια ποσότητα, ένα νούμερο το οποίο αν το διαιρέσουμε δια του αριθμού των κρατών μελών είναι ψίχουλα για το κάθε κράτος μέλος για κάθε κράτος μέλος λοιπόν η συνεισφορά δεν τη νιώθει, δεν το τσούζει όμως συνολικά αυτή η πόρη είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και δίνει τρομακτική προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο ελπίζω ότι θα είμαστε όλοι σύμφωνοι τελικά και ότι θα θελήσουν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την προτάσή μας. Είμαι πεπισμένος, επαναλαμβάνω, τα 280 εκατομμύρια ευρώ με νέο χρήμα και με το εργαλείο ευελιξίας χωρίς να έχουμε εκ νέου διοχέτευση από παλαιότερα ε, κονδύλια είναι κάτι το εφικτό. Καταληκτική προθεσμία 27 Μαρτίου για τις τροπολογίες. Αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα το ψηφίσουμε στις 16-17 Μαΐου στην Επιτροπή μας και ε, στην Ολομέλεια του Ιουλίου στη συνέχεια. Και ελπίζω ότι στην Ολομέλεια θα εγκριθεί ε, το κείμενο και θα μπορέσει να ληφθεί η απόφαση το γρηγορότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και να σας ε, επισημάνω ότι η γραμματεία μας σήμερα το απόγευμα θα αποστείλω την υποποιημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας πω ότι άλλαξε και η αριθμίση των παραγράφων και ως εκ τούτου πεστάλλει ένα αντραστικό σημείωμα. Σας παρακαλώ λοιπόν στις τροπολογίες να λάβετε υπόψη αυτή την αλλαγή της αριθμίσης γιατί ιδάλλως θα προκληθεί σύγχυση. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διατάξη. Η αποστολή στην Ιρλανδία 12 μέχρι 14 Φεβρουαρίου του 2018 και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Ρούμπιχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την γραμματεία όλους ιδιαίτερους για την προετοιμασία της αποστολής αυτής στην Ιρλανδία ήταν καθοριστική σημασία. Το ότι λάβαμε την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γεγονός ότι έγινε μια συζήτηση με τους πολίτες, με ΜΚΟ, με επιχειρήσει, με εταιρείε και υπό την παρουσία του Δημάρχου του Δουβλίνου, ακαδημαϊκών κύκλων. Ε, επίσης συναντηθήκαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπου είδαμε τι επιδόσει και τη Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, με τον Υπουργό ε, Προπολογισμού, ε, με τον επικεφαλής της Επιτροπή Προπολογισμών. Επισκεφτήκαμε διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι και η Ιρλανδία στο πλαίσιο του πολιτές δημοσιονομικού πλαισίου έχει ξεκινήσει σημαντικές συζητήσει σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, σε ό,τι αφορά την ΚΑΠΑ, αποτελούν τι παραδοσιακέ αν θέλετε, τα παραδοσιακά ζητήματα, αλλά και το Erasmus Plus και η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν ζητήματα και τα νέα μέσα τα οποία θα προβλεφθούν στον προπολογισμό και το πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία στον τομέα της άμυνας, τι γίνεται με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι τα σημεία επικέντρωση σε ό,τι αφορά το κυβέρνο έγκλημα τη ψευδή ειδήσει, τα συνηθισμένα ζητήματα. Το Brexit δεν ήταν επίσημο θέμα, αλλά όταν μιλάμε φυσικά για πολύ δημοσιονομικό πλαίσιο, πάντα ανακύπτει το θέμα αυτό. Ήταν αισιόδοξε ωστόσο οι προβλέψει. Η βασική εταίροι ε, έχουν ε, αρκετά αισιόδοξη προοπτική σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία αποχώρηση, τι μεταβατικέ ρυθμίσει κτλ. γίνονται κάποιες προετοιμασίες για το τι θα γίνει σε περίπτωση σκληρού Brexit, αλλά δεν θεωρείται πιθανό αυτό. Ανέκυψε και το ζήτημα των εσωτερικών πολιτικών ζητημάτων της, στον Βασίλειο σε ό,τι αφορά την τοποθετήση της Ιρλανδίας, της Σκοτίας και του Γεβραλτάρ που θα ήταν υπέρ της παραμονής στην Ένωση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα τεθεί θέμα συνόρων. Νομίζω ότι θα έχουμε και Προφανώ εξασφαλισμένο μέλλον σε ό,τι αφορά την ενεργειακή συνεργασία. Γενικά ήταν λοιπόν θετικό το κλίμα και δεν γίνεται προετοιμασίε, θα έλεγα, για ένα σκληρό Brexit. Μα ζητήθηκε να προετοιμάσουμε και ένα σενάριο σε περίπτωση που μία από τις τρεις βουλές δεν συνενέσει, δεν συγκαταθέσει, δώσει συγκατάθεση για τη συνθήκη αποχώρηση και το πώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί η κατάσταση σε περίπτωση τέτοια για τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά γενικά ήταν θετικό το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο, η συνάδελφο Νιρήρα. Um, ευχαριστώ τη Γραμματεία για την διοργάνωση και ήταν πολύ ωραίο που πήγαμε μαζί με τους συναδέλφους επί Έχω ε, μια, κάνω κάποιες διαφορετικές σκέψεις. Ε, όταν μιλάμε για το Brexit δεν νομίζω ότι υπάρχει αισιοδοξία ε, γι' αυτό. Ε, όταν ο κόσμος μιλάει μεταξύ του ε, υπάρχει συνειδητοποίηση ότι το θέμα δεν είναι μόνο θέμα συνόρων, θα επηρεάσει ολόκληρη την Ιρλανδία. Νομίζω ήταν σημαντικό η Επιτροπή Μπάτζ να δει τι λέει ε, ο Ιρλανδικό Λαό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πά στην Ιρλανδία για να, και να γνωρίσει το θέμα του Brexit, γιατί θα μας επηρεάσει παντού, ε, βορρά, νότο, ανατολή, δύση του νησιού. Ήταν πολύ επωφελές λοιπόν για του Ιρλανδού να δουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τους αντιμετωπίζει σοβαρά ε, όσο ό,τι αφορά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πώς επωφελούμαστε κτλ. Και τι συμβαίνει όταν στερέψει αυτή η πηγή. Η έκθεση είναι καλή, Ευχαριστώ τους συναδέλφου και ειδικά τη γραμματεία που έκανε τόσο καλή δουλειά. Πρέπει να ξανάρθει του χρόνου. Μετά τις εκλογές βέβαια. Ναι. Βεβαίω, πολύ θα ήθελα κι εγώ, γιατί φέτο δεν μπόρεσα να συμμετάσχω και θα ήθελα πολύ να ξαναπάω. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώσαμε σχεδόν ε, το, την ημερήσια διάταξη. Να σα επισημάνω το εξή στι 16 Απριλίου, τη Δευτέρα απόγευμα, στο Στρασβούργο θα πρέπει να συζητήσουμε τις προθεσμίες για τον ε, προπολογισμό του Κοινοβουλίου προκειμένου να τα λάβει υπόψη αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας είναι εδώ στις Βρυξέλλες ε, στις 23 και 24 Απριλίου. Και έτσι λοιπόν λέει τη συνεδρίαση.